Συνάδελφοι. Can Λοιπόν, έχουμε την ομάδα κρούσια του τουρισμού. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, να ηρεμήσουμε και να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα θα συζητήσουμε το έγγραφο εργασία τοποθέτηση. όσον αφορά τη διάσκεψη για την κληρονομία του τουρισμού που θα γίνει 25 Απριλίου στο Δουβλίνο γιατί έχει καθυστερήσει ο Επίτροπο Ταγιάννη. Ο Κάρλο Φιντάνσα θα προεδρεύσει όταν έρθει και ο Ταγιάννη. Η Κάρλα μάλλον γιατί έχω άλλη... έχω να πάω στο γιατρό και θα πρέπει να φύγω. Πάμε λοιπόν στη διάσκεψη για την ε, τουρισμό, για την κληρονομία στον τομέα του τουρισμού στο Δουβλίνο, 25 Απριλίου. Θα έχετε ένα έγγραφο λοιπόν στο φάκελό σας που συνέταξε αυτή η ομάδα κρούσης Προτείνω να καθορίσουμε προθεσμία 14 Απριλίου 12 το μεσημέρι για όποιον θέλει να προσθεθεί κάτι στο συγκεκριμένο έγγραφο. Θεωρήσαμε ότι θα είναι καλό να έχουμε αυτό το έγγραφο τοποθέτησης για αυτή τη διάσκεψη και ελπίζουμε να βοηθήσει, να συνεισφέρει στις συζητήσεις. Τους λέμε κάποια πράγματα για μας. Αναφέρουμε και τις προτεραιότητές μας. Προτεραιότητες που συμπεριλαμβάνονται σε διάφορες ε, εκθέσεις μας. Αναφέρεται και στις ε, μελέτες που έχουμε ετοιμάσει. Δεν ξέρω για την ώρα κατά πόσο εγώ, ο Κάρλο ή κάποιος από τους ε, αντιπροέδρους θα είναι παρόν στη διάσκεψη. Δεν έχουμε προσκληθεί επίσημα. Αν ξέρει κανείς ποιος στέλνει τις επίσημες προσκλήσεις, σας κάνει κάτι να προσθεθούμε στον κατάλογο. Θεώρησα όμως ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε την περίσταση για να υποβάλουμε αυτό το έγγραφο με τις θέσεις μας. Μέχρι 14 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι μπορείτε να στήσει να προσθεθεί κάτι κλπ. Έχετε κάποιες ερωτήσεις. Κάρλο, θες να προσθέσεις κάτι. Ευχαριστώ Μπράιον. Προτείνω να μιλήσει ο συνάδελφος Higgins για την επίσημη πρόσκληση, πέρα λοιπόν από τα αστιάκια, είναι σημαντικό η Task Force και η Επιτροπή να είναι παρούσα σε αυτή τη διάσκεψη της Ιταλικής Προεδρίας με μια τοποθέτηση πάνω σε ένα θέμα στο οποίο εξάλλου επανειλημμένα έχουμε τοποθετηθεί και υπενθυμίζω και εγώ και οι συνάδελφοι για δεύτερη συνεχή χρονιά θέλουμε να διατεθεί ένα ποσό στον προπολογισμό της, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του προπολογισμού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δοθεί ένα κονδύλι για να αναπτυχθούν διάφορα προγράμματα όσον αφορά τον πολιτισμικό τουρισμό, την αξιοποίηση ε, της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Είναι σημαντικό θέμα και θα πρέπει να δοθεί συνέχεια σε αυτή την προσπάθεια. Να είμαστε παρόντες λοιπόν σε αυτή τη διάσκεψη σε μια, με μια τοποθέτηση. Και εγώ έχω λάβει το έγγραφο αυτό μόλις τώρα, οπότε επιφυλάσσομαι για ε, παρατηρήσεις, ε, τυχόν, προτάσεις για προσθήκες στο κείμενο. Εντός της προθεσμίας που έχει προβλεφθεί εντάξει, ικανοποιημένη, 14 Απριλίου είναι η προθεσμία. Ο Κιθ, ευχαριστώ Μπραέν. Ρώτησες κατά πόσο έχουμε ερωτήσεις, έτσι. Όχι, δεν έχω ερωτήσεις και δεν είμαι σίγουρος αν είναι η σωστή στιγμή να το αναφέρω αυτό ή η επόμενη συνεδρίαση της Task Force ίσως θα έπρεπε να το ζητήσει. Και α, το θέμα, η ευημερία των ζώων και η προστασία των ζώων στη, στον τουρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θυμόσαστε ότι η Ένωση ε, των Βρετανών αρμοδίων για το θέμα Έδωσε κατευθυντήριες γραμμές λοιπόν στον τομέα του τουρισμού για την επιμερία των ζώων και είχε εκδοθεί έκθεση πέρσι και είχε πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα προωθούσε τις κατευθυντήριες γραμμές αυτής της οργάνωσης της ΑΠΤΑ και θα τις υιοθετούσε. Νομίζω ότι είναι ένα αρκετά καλό μήνυμα, ώστε η ευημερία των ζώων να μπει σαν μία ακόμη προτεραιότητα στο σχέδιο εγγράφου τοποθέτησης ή και να επανέλθει σε αυτή την ε, ομάδα κρούσης για τον τουρισμό, στην Task Force. Ε, υπάρχουν αντιδράσεις. Εγώ θα έλεγα, Keith, για όσο αξίζει η γνώμη μου, συζητήσουμε το θέμα της ευημερίας των ζών στον τουρισμό της υπαίθρους. Μπορεί αυτό να μπει σαν θέμα για μελλοντική συνάντηση της ε, Task Force αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι όταν επανέλθουμε μετά το Πάσχα μαζί με τον Κάρλο να προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε τα θέματα που θα συζητήσουμε και πώς θα τα συζητήσουμε. Ε, πρόθεσή μου λοιπόν είναι αυτό να το κάνουμε μετά το Πάσχα μαζί με τον Κάρλο και ένα από τα θέματα προς συμπερίληψη θα μπορούσε να είναι και αυτό η ευημερία των ζώων. Μπορεί να μας στείλει ένα email με αυτή την πρόταση για να τη δω στο χαρτί μπροστά μου και μην την ξεχάσω ε, όσον αφορά το πακέτο για τον σιδηρόδρομο, για, ε, για πτήση, ώρα υπηρεσίας κλπ. κλπ. Όλα αυτά τα θέματα. Θα το λάβουμε υπόψη και ο Κάρλο και εγώ, όπως προανέφερα, μετά το Πάσχα θα προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε το πώς θα προχωρήσουμε με αυτή την ομάδα του τουρισμού. Ξέρω ότι και ο Κάρλο έχει κάποιε ιδέε, θα τι εξετάσουμε και θα το κουβεντιάσουμε. Καλώ. Είστε όλοι ικανοποιημένοι. Ωραία. Περιμένουμε για τον Επίτροπο. Πόσο χρόνο χρειάζεται, ξέρουμε. Έχουμε μια ιδέα. Θα πρέπει να, να καταφτάσει όπου να είναι. Οπότε μπορούμε έτσι να αλλάξουμε και τα πινακάκια και να έρθει να καθίσει εδώ ο Καρλός στη μεγάλη καρέκλα. Λοιπόν, λίγη υπομονή να περιμένουμε για την αύξηση του Επιτρόπου. Bene, riprendiamo i nostri... Καλώς. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Καλώς ορίζουμε τον Τριπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αντώνιο Ταγιάννη που κατέφθασε. Θέλαμε πολύ να έχουμε αυτή τη συνάντηση για λόγους ε, φορτωμένου χρονοδιαγράμματος του Αντιπροέδρου από τη μία και των δικών μας εργασιών από την άλλη δεν καταφέραμε να οργανώσουμε αυτή τη συνάντηση πιο νωρίς και αυτό εν μέρη καθυστέρησε και τις εργασίες ε, της Task Force μας, αλλά πιστεύω ότι είναι θεμελιώδου σημασία να γνωρίζουμε εμεί ε, ακριβώ σε ποιο στάδιο έχουν φτάσει οι δραστηριότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για διάφορα κεφάλαια τα οποία μα απασχολούν και τα θεωρούμε ως προτεραιότητε όσον αφορά την πολιτική του τουρισμού. Δηλαδή τη δουλειά που κάνουμε στο Κοινοβούλιο και στην έκθεση που ενεκρίθη τον Οκτώβριο 2011 και με τη δημιουργία της ομάδας κρούσης και με το έγγραφο με τις προτεραιότητες που, ετοιμάσαμε, που ξεκινήσαμε να ετοιμάζουμε εδώ και μερικούς μήνες. Δηλαδή μια ενημέρωση όσον αφορά τα διάφορα θέματα θα μπορεί να μας δώσει τώρα και ο Αντιπρόεδρος και είναι θεμελιώδες αυτό και για να αναπρογραμματίσουμε αν θέλετε ε, και τις δράσεις μας, λεπτομέρειες των δραστηριοτήτων μας βάσει των προτεραιοτήτων που έχω θέσει χωρίς να καθυστερώ Δίνω το μικρόφωνο στον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Ταγιάννη. Ευχαριστώ, αγαπητέ Κάρλο, ευχαριστώ όλους σας. Έφτασα κάπως καθυστερημένα, διότι συμμετείχα στο φόρουμ για το Δούναβι, στη διάσκεψη για το φόρουμ του Δούναβι, της, που διοργάνωσε η κυρία Τικάου. Είχα υποχρέωση λοιπόν. Και έχουμε και την κοιλάδα του Ταγιάννου κοντά αφορά την Ισπανία, Ρουμανία και ο Ταϊανός ήταν ε, ο πρώτος αυτοκάτος, μπορέσαμε να βρούμε και συσχετισμούς μεταξύ Δύσης, Ανατολής και λοιπά της Ευρώπης. Ο τουρισμός είναι σημαντικός και γι' αυτό, διότι έτσι γνωρίζουμε καλύτερα ένα τον άλλον, επιτρέπει να αξιοποιούμε τις κοινέ μας ε, ρίζες, αλλά είναι και ένα έξοχο εργαλείο για την οικονομία μας. Για πολύ καιρό ο τουρισμός ε, θεωρείται ένα είδος ταχτοπούτας όσον αφορά την οικονομική μας ε, πολιτική. Ευτυχώς η συνθήκη της Λισαβόνας έδωσε νομική βάση για μια ευρωπαϊκή πολιτική τουρισμού που δεν θα πρέπει να παραβιάσει επουδενή την αρχή της επικουρικότητας αλλά θα πρέπει να δίνει προστιθέμενη αξία. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους αξιότιμους κυρίους Σίμψον και Φιντάνς που θέλησαν να υποστηρίξουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την έκθεση του 2011 που έριξε την ιδέα της δημιουργίας της Task Force της ομάδας κρούσης που κατά την άποψή μου εργάζεται με πολύ θετικό τρόπο. Είναι σημαντικό να υπάρξει ένα συντονισμός των δράσεών μας 21 προτάσεις είχαμε κάνει. Εργαζόμαστε πολύ όσον αφορά τουλάχιστον την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υλοποιήσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει και τις προτεραιότητες. Και αυτό επειδή διότι μπορώ να υποστηρίξω στην πολύ στεναρή υποστήριξη του Κοινοβουλίου και θα ήθελα να ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω πάνω απ' όλα για την υποστήριξη που μας δόθηκε που προβλέπει και παρεμβάσεις ε, υπέρ του τουρισμού η τοποθέτηση. Θα έλεγα ότι αναγνώρισαν πάντες και μέσω των δράσεων της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανακοινώσεων Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναγνώρισαν όλοι ότι τα πράγματα αλλάζουν και πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο τουρισμός είναι ένας τομέας οικονομικός και μπορούμε πραγματικά να, τον, να βάλουμε στην πρώτη γραμμή τον τουρισμό σαν δράση κατά της κρίσεως και για τη θέση, απασχόλη, θέση απασχόλησης. Όπως ξέρετε, είναι ο τομέας στον οποίο απασχολούνται περισσότεροι νέοι και, ε, και δημιουργεί 100.000 θέσεις εργασίας το χρόνο. Ε, και ο τουρισμός μπορεί να διαδραματίσει μεγάλο αλληλοεπηρεάζει την, την, ε, ε, το ζήτημα της ε, εποχικότητας και νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να αναφερθώ στο ότι μπορούμε να υιοθετήσουμε και στο θαλάσσιο τουρισμό προγράμματα επιτυχημένα στον, σε άλλες μορφές τουρισμού όπως ήταν το ίντεν ή το καλύψο που, σήμερα μέχρι σήμερα δεν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε στο θαλάσσιο τουρισμό. Τέλος, σε σχέση με την κουραζιέρα που είναι μια αναπτυσσόμενη μορφή θεματικού τουρισμού με εξαιρετικές υποσχέσεις ε, για την Ευρώπη. Ε, νομίζω ότι ε, βασικό ζήτημα, θέμα κλειδί για να μπορέσουν τα, τα λιμάνια να γίνουν λιμάνια port homes και όχι διέλευσης, που αυτό είναι βεβαίως το ζητούμενο, πρέπει να αντιμετωπιστούν μια σειρά αποζητήματα πέρα από τα τεχνικά και τα ζητήματα υποδομής που έχουν να κάνουν και με το θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε λίγο πριν με την πολιτική των της βίζας, των θεωρήσεων βίζα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Ε, κλείνοντας, νομίζω ότι η, η ομάδα μας ε, μέσα σε ένα ε, συνεκτικό προγραμματισμό δράσεων ε, που έχει καταρτήσει εκτιμά ότι θα σας έχει σταθερό σύμμαχο και συνεργάτη γιατί και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα, ιδιαίτερα σε αυτήν την δύσκολη συγκυρία, όπως είπαμε και πριν, ε, του τομέα του τουρισμού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, De Grandes και μετά Higgins. Sí, muchas gracias, señor. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φιντάν. Θα θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο και Επίτροπο Ταγιάννη Αργήσατε να φτάσετε, αλλά πάντως φτάσατε έγκαιρα. Και η Κομισιόν και η Ευρώπη ε, είναι τυχερή που έχει εσάς να ασχολείστε με αυτό το θέμα πραγματικά. Διότι κάποιες φορές ο τουρισμό θεωρείται εξωγενή τομέα σε ό,τι αφορά την οικονομική δραστηριότητα σε κάποιες χώρες, Όχι όμως για τη δική μου χώρα είναι ένας από του σημαντικότερους τομεί ε, μια από τις σημαντικότερες ε, βιομηχανίες. Ε, η πολιτική τώρα συνεργασία, ανταλλαγή, πολιτισμική, η Task Force και όλα αυτά τα συζητήσαμε και είναι γεγονός ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση στον τουρισμό ως πηγή πλούτου και είναι μια καλή ιδέα αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει να σας συγχαρούμε γιατί πραγματικά κινείστε σε λεπτά σε ένα έδαφος δύσκολο. Έχουμε το άρθρο 195 της συνθήκης εναρμόνισης, ε, αλλαγή και μια ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική που σέβεται και την αρχή της επικουρικότητας. Όλα αυτά πρέπει να τα συνδυάσετε. Ο Κάρλο Φιντάντσα ο πρόεδρος της Task Force, συμμετέχω και εγώ. Συμφωνώ με όσα είπατε από το Α στο Ω, αλλά θέλω να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση ε, με όσα είπατε κάτι πρέπει να γίνει με κάποιους τουρίστες. Είναι μια ε, πάρα πολύ καλή ιδέα σε ό,τι αφορά τη θεώρηση διαβατήριων Κινέζων ε, τουρισμών, τουριστών. Ευτυχώς ε, στην Κίνα δεν ισχύει ότι στην Κούβα, παρότι υπάρχει κομμουνιστικό καθεστώς, επιτρέπεται στους Κινέζους να φεύγουν από τη χώρα, να επισκέπτονται άλλες χώρες και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πλούτο για τη δική μα Ήπειρο. Έχουμε όμως ένα εκκρεμέ ζήτημα με τις ΗΠΑ. Ε, οι Αμερικάνοι δεν έρχονται ε, στην Ευρώπη. Έχουμε πολύ χαμηλά επίπεδα ε, παρουσίας, προσέλευση Αμερικανών τουριστών στην Ευρώπη. Και υπάρχουν κάποια άλλες χώρες του Βορρά που ναι μεν αυξάνουν τις τουριστικές ροές, αλλά αυτό που παρατηρούμε είναι το αντίστροφο κυρίως, δηλαδή ότι άνθρωποι από τον νότο πηγαίνουν όλο και περισσότερο προς το βόρειο και όχι το αντίστροφο. Ίσως η κρίση, πάντως πρέπει να αυξηθεί, δεν πρέπει να δώσουμε έμφαση στην αύξηση τουριστικών ροών από τις ΗΠΑ. Τώρα η ποιότητα δεν πρέπει να μείνει στα λόγια, πρέπει να γίνει μια πραγματικότητα και θα σας δώσω και κάποια στοιχεία Μέχρι το Φεβρουάριο χάσαμε 1,3% ε, ενώ αυξήσαμε κατά 5,1% σε δαπάνες. Δηλαδή η ποιοτική προσφορά ε, μπορεί να δώσει θετικά αποτελέσματα. Η Ρώσα Εσταράς, η Νέσα Γιάλα έχουν πολλές φορές πει η πρώτη βέβαια δεν συμμετέχει στην αλλά μα δίνει την εμπειρία από τη Μαγιόρκα. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να λάβουμε υπόψη μα είναι ο κοινωνικό τουρισμό, ο λεγόμενο. Senior. Δυστυχώ ε, μειώνονται οι γεννήσει, αυξάνονται οι ηλικιωμένοι σε σχέση με του νέου. Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στους, στην τρίτη ηλικία, στους συνταξιούχους, να μπορούν και αυτοί να ταξιδεύουν περισσότερο ή να εκμεταλλευόμαστε κάποιε νεκρέ εποχέ για τα ξενοδοχεία, για παράδειγμα, να ταξιδεύουν τότε. Και το καλυψό είναι κάτι το οποίο θέλω να επικροτήσουμε. Τώρα, και ο νεανικό τουρισμό είναι κάτι που πρέπει να στηρίξουμε. Σήμερα στα πρωτοσέλιδα σχεδόν των μέσων ενημέρωση στην ε, Ισπανία λέει ότι αυτά τα πακέτα νέων, ε, αν μπορεί να τα πει κανείς πακέτα, τέλος πάντων νέοι οι οποίοι ε, ταξιδεύουν ότι δεν είναι κάτι το ευκταίο. Ε, το μόνο που κάνουν, παραδείγματος χάρη όταν πηγαίνουν να συμμετάσχουν σε μια αθλητική διοργάνωση να δουν, το μόνο που κάνουν είναι να τα πίνουν. Δηλαδή δεν πάνε ούτε καν στο στάδιο ή κάπου που εξάγεται μια αθλητική εκδήλωση, αλλά πάνε σε ένα μπαρ και μένουν εκεί πέρα. Το θέμα είναι να δούμε αν μπορούμε να βοηθήσουμε με εκπαιδευτικά προγράμματα. Πρέπει να προσέξουμε. Βέβαια δεν φταίει η Ευρώπη γι' αυτό ε, όλοι μας στις χώρες μας πρέπει να προσέξουμε τι γίνεται με τέτοιου είδους ε, ταξίδια ε, νεολαίων. Τώρα αυτά τα 231 εκατομμύρια είναι πολύ καλοδεχούμενα. Τώρα πρέπει να δούμε κατά πόσον θα αποδειχθεί τελικά και όταν αποδειχθεί ότι είναι πηγή ελπίδας και πλούτο τουρισμός για όλους μας, μήπως τότε όταν αποδειχθεί αυτό να ε, ληφθούν υπόψη και οι χρηματοοικονομικές ανησυχίες που δεν είναι έλασον αλλά μείζον ζήτημα. Υπάρχουν χώρες που νόμιζαν ότι δεν είχαν τις δυνατότητες ε, αλλά τις έχουν και για να υποδέχονται κόσμο αλλά και για να στέλνουν κόσμο προς τα έξω. Είναι μια επιτυχημένη ε, ιστορία κύριε Επίτροπε, είναι μια επιτυχία που έχουμε να προβάλλουμε και είναι θετικό για όλους μας. Ευχαριστώ. Grazie. Higgins e poi Estaras. Ευχαριστώ, Higgins. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να πω πως συμφωνώ με τον Αντιπρόεδρο πως ο τουρισμός ήταν η στεφτοπούδα. Η επιτροπή μας ήταν η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού και μέχρι ο Κάρλο Φιντάντσα να παρουσιάσει ένα σχέδιο έκθεσης με τίτλο Ευρώπη, ο πρώτος ε, τουριστικός ε, προορισμός του κόσμου, δεν μιλούσαμε για τον τουρισμό. Είναι λοιπόν καλό το έγγραφο. Το πρόβλημα που έχουμε τώρα είναι το εξή. Κύριε Αντιπρόεδρε, μιλάμε με γενικότητες. Δεν έχουμε συγκεκριμένους στόχους, έχουμε έναν προπολογισμό πολύ μικρό, αλλά είναι μία αρχή. Μιλάμε για εποχικότητα και αυτό είναι όλο. Μιλάμε για τον ιστορικό τουρισμό και τέλος. Δεν έχουμε κάποιο σχέδιο για το προς τα που θέλουμε να πάμε, να κινηθούμε. Οπότε χρειαζόμαστε στόχους, πιο συγκεκριμένα πράγματα δηλαδή. Και θα έλεγα και το εξής. Σας ακούω. Και ο συνάλφος ο Λούς το ανέφερε και το αναφέρετε και εσείς κύριε Πρόεδρε όσον αφορά τη σήμανση ποιότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να ξέρει ο κόσμος τι ε, αγοράζει όταν αγοράζει ένα προϊόν. Τι είδους ε, στέγη, τι φαγητό, τι αξιοθέατα υπάρχουν κτλ. Εσείς είπατε πως σκοπεύετε να έχετε ένα έγγραφο του επόμενου μήνες. Έχω ένα πρόβλημα εδώ πέρα, γιατί όταν ακούω την Κομισιόν να λέει τους επόμενους μήνες, σημαίνει τα επόμενα χρόνια στην πράξη. Οπότε, έχετε συγκεκριμένη προθεσμία συγκεκριμένη ημερομηνία. Δεύτερον, θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν να μας πει τι χρήματα, ξέρω πως ο προπολισμός είναι μικρός, αλλά μιλάμε για πρόθεση της Ευρώπης σε Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα. Έχετε ορίσει προπολογισμό για αυτές τις τέσσερις χώρες, γιατί είναι ο στόχος μας. Η Βραζιλία, Κίνα, Ρωσία και Ινδία. Πρέπει να τα ξέρουμε αυτά. Τρίτον, σε σχέση με την οδηγία των ταξιδιωτικών πακέτων από το 1990 πρέπει να αναθεωρηθεί επιτέλους. Πότε θα αναθεωρηθεί. Είναι πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις, αλλά έτσι κάνουμε στην Ιρλανδία. Και τέλος πρέπει να σκεφτούμε και με τρόπο πρωτότυπο. Εμείς εξαρτώμεθα 35% της οικονομίας μας από τον τουρισμό. Επειδή λοιπόν υπάρχει ένας ε, τεράστιος αριθμός ε, ανθρώπων που έχουν Ιρλανδικές ρίζες, μεταξύ των οποίων, κάτι 17 εκατομμύρια άνθρωποι, μεταξύ οποίων και ο, ο Ομπάμα, τους ε, λέμε να έρθουν στην ε, Ιρλανδία, να βρουν που γεννήθηκε ο προπάπους τους. Ε, και Έχουμε βεβαίω και ειδικά πακέτα, πτήσεις και ελπίζουμε πως όταν έρθουν μια φορά θα ξανάρθουν. Κυρίως από τις ΙΠΑ στην Ιρλανδία. Και τέλος η απαλλαγή βίζας. Πρέπει να γίνει κάτι με αυτό. Το αναφέρατε κι εσείς. Πότε όμως. Ε, αυτό είναι το ερώτημα. Σας ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Σα Σας ευχαριστώ, Εστεράς και τα ξέρω. Ε, ευχαριστώ κύριε Φιντάτσα. Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ τον Επίτροπο για το έργο του. Τον συνάδελφο βέβαια Κάρλο Φιντάντσα και τα μέλη της Επιτροπής μας και ιδίως τον σύντροφο Λουίς Ντεγκράντες που ασχολείται με όλα αυτά τα ζητήματα του τουρισμού εξαιρετικό τρόπο. Έχω να κάνω δύο-τρία σχόλια. Εποχικότητα, είπε και ο Επίτροπος, είναι πάρα πολύ σημαντικό να την καταπολεμήσουμε γιατί περισσότερες τουριστικές οικονομίες στην Ευρώπη είναι εποχικές. Άρα εναλλακτικό τουρισμός ε, σε όλες τις μορφές θα πρέπει να μελετηθεί εμπορικός, ε, υγείας, ε, εινοποιίας, ο ιστορικός και κτλ. λοιπά. Έπειτα η εκπαίδευση και η αριστεία στην εκπαίδευση είναι πάρα πολύ, θα θεμελιώδης ε, πτυχή και έπειτα συμπληρωματική προσφορά. τι μπορούμε να προσφέρουμε στα τουριστικά πακέτα. Τώρα η αριστεία, είπα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και για την έρευνα και ανάπτυξη, γιατί τα τουριστικά πακέτα αγοράζονται με διαφορετικό τρόπο. Σε πολύ μεγάλο βαθμό γίνονται online από εταιρείε ε, οι οποίε έχουν ε, εισχωρήσει στην αγορά και πρέπει να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Το σημείο κλειδί όμω είναι ποιότητα και διασύνδεση. Δεν μπορούμε να ε, είμαστε ο πρώτο τουριστικό προορισμό αν δεν έχουμε διασύνδεση, δυνατότητα διασύνδεση. Πάρα πολύ καλά τα είπε ο κύριο Λίς Δεγκράντες, πράγματι προσωπώ τη Μαγιόρκα και είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μπορούμε να έχουμε διασύνδεση Δηλαδή κυρίω ε, να έχουμε παραδείγματο χάρη ε, με τις εταιρείε, με τις πτήσει ε, διασύνδεση. Έχουμε α πούμε απευθεία πτήση από την Πετρούπολη το Σεν Είναι σημαντικό να υπάρχουν αεροπορικές συνδέσεις, ιδίως με τα νησιά. Αλλά και από και προς ε, τους βασικότερους προσμούς στην Ευρώπη. Επίσης, Θέλουμε να προωθήσουμε την υπεύθυνη ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα. Άρα, οπωσδήποτε πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ποιότητα. Η ποιότητα στον τουρισμό είναι σαν να μιλάμε για βιώσιμο περιβάλλον, για εφόρο περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντική ποιότητα και σημαίνει και περισσότερη ανταγωνιστικότητα, μεγαλύτερη οικονομική πρόοδο. Και γι' αυτό θέλω να επικροτήσω και την πρωτοβουλία του Επιτρόπου που ανεστά αυτή την εναρμόνιση και όταν έχουμε αυτό το σήμα ποιότητας ε, πρέπει να δώσετε έμφαση σε αυτό γιατί έχουμε σήματα, πολλά σήματα, αλλά όχι ένα σήμα ποιότητας, σε τίποτα ουσιαστικά. Ούτε στην ποιότητα της συμπληρωματικής προσφοράς, ούτε των ξενοδοχείων, της ξενοδοχής προσφοράς. Θα πρέπει να μιλήσουμε και για την προσπελασιμότητα, την προσβασιμότητα. Έχουμε 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία στην Ευρώπη. Αν θέλουμε να έχουμε μια ε, Ευρώπη που να προσφέρει ισότητα ε, στι αξίε και ισότιμε ευκαιρίε, η αναψυχή, ο τουρισμό και εκεί πρέπει να εξασφαλίζεται αυτή η ισότιμη πρόσβαση και για τα άτομα με αναπηρία όχι μόνο όμως από αυτή την πτυχή της αναπηρίας, αλλά και από την πτυχή της ποιότητας. Πώς θα προσελκύσουμε αυτά τα 80 εκατομμύρια ατόμων με αναπηρία. Επίσης έχουμε πάνω από 20 διαφορετικά λογότυπα για να δούμε αν είναι προσβάσιμος ή όχι ένας προορισμός. Ασφάλεια και προσβασιμότητα είναι το πρώτο. Αλλά δεν είναι ο ίδιος λογότυπος ε, σε κανένα σχεδόν κράτος μέλος. Άρα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να κάνουμε μία μεγενοποίηση ε, των λογοτύπων. Και τέλος, ε, θέλω να πω ότι ο τουρισμός είναι ένα εγκάρσιο ε, θέμα. Τι εννοώ με αυτό. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Θόρυβος. Μπορεί να γίνονται έργα σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων ή τεσσάρων όταν τότε είναι η high season λεγόμενη ε, όταν ε, είναι περίοδος διακοπών. Μα δεν μπορεί ένας τουρίστα να ακούει κομπρεσέρ ε, συνέχεια. Τι πρέπει να κάνουμε με αυτό το θέμα, με το θέμα της χορύπανση, γιατί πραγματικά επηρεάζει πάρα πολύ τον τουρισμό. Πρέπει να τηρούνται αυτέ οι παράμετροι ποιότητα, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι διαφορετικέ ρυθμίσει που ισχύουν σε κάθε κράτο μέλο. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν, γιατί μας το ζητάει και η Ισπανική Ομοσπονδία Ξενοδοχείων, αν μπορούμε να έχουμε ένα πλαίσιο Βέβαια υπάρχει αρχή της επικουρικότητας, αλλά τέλος πάντων αυτά τα εγκάσια θέματα πρέπει να ρυθμιστούν. Ή τα δικαιώματα δημιουργού, πραγματικά δικαιώματα. Μπορεί αυτό να επηρεάσει όταν τα ξενοδοχεία, για παράδειγμα, πρέπει για τις ε, τηλεοράσεις, για παράδειγμα, τι γίνεται. Ακόμη και όταν μπορεί να είναι κλειστά ε, για κάποιο διάστημα, αλλά πρέπει να πληρώνουν κάποια δικαιώματα. Αυτά είχα να πω και θέλω να ευχαριστήσω και τον Κάρλο Φιντάντς. Ε, σε ευχαριστώ Ρόζα. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσω ότι δεν θα δώσω του λόγου σε εναλλαγή πολιτικών ομάδων. Θα το καταλάβατε. Ακολουθούμε σειρά, με τη σειρά που ζητήσατε το λόγο. Γι' αυτό δεν ήταν θελήμα μίλησαν διάφοροι του ΕΛΚ, απλώ ήταν η σειρά που είχαν ζητήσει το λόγο. Θα παρακαλούσα του συναδέλφου που θα μιλήσουν σύντομα να είναι λίγο πιο λακωνική για να δώσουμε τη δυνατότητα στον Αντιπρόεδρο να απαντήσει σε όλες τις σωστές ερωτήσεις που θέτεται. Τεξέρα και Φώστερ. Ευχαριστώ. Και Επιτροπέ, σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα να μας ε, μιλήσετε και είστε στη διάθεση της Επιτροπής μας. Επίσης να συγχαρώ τον Καρλ Φιντάντσα για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία για μια ομάδα εργασία για τον τουρισμό που μπορεί νομίζω στο μέλλον να συνεισφέρει σε μια πραγματική ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα εμβριακό στάδιο. Αναφέρατε τη σημασία του τουρισμού για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Πορτογαλία είναι γύρω στο 11% του ΑΕΠ μας και γύρω στο 12% των θέσεων εργασίας. Εγώ λοιπόν Προέρχομαι από μια απομακρυσμένη περιοχή και εκεί πέρα ο τουρισμός είναι γύρω στο 30% της τοπικής οικονομίας. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντικός είναι για εμάς. Τώρα. Αναφέρεται κάποιες προτάσεις ε, για την ομάδα εργασίας και υπάρχουν δύο προτάσεις που νομίζω πως πρέπει να εξετάσουμε πρώτα απ' όλα μια ομάδα διαχείρισης της κρίσης για τον τουρισμό. Όλοι γνωρίζουμε το πόσο έχουν τις δυνατότητες να ε, επηρεάσουν τον τουρισμό φυσικές ε, καταστροφές. Ε, στη Μαδέρα το 2010 είχαμε μια φυσική καταστροφή, λάβαμε και βοήθεια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης και τις μέρες μετά την 20η Φεβρουαρίου είχαμε 10.000 ακυρώσεις και βεβαίως αυτό είχε φοβερό αντίκτυπο. Πρέπει κανείς μετά βεβαίως και να καθαρίσει την περιοχή κτλ. Αλλά δεν γίνεται καμία προσπάθεια για να ε, αποκατασταθεί η ροή η τουριστική. Αυτό πρέπει να δούμε. Μία άλλη πρόταση για την ομάδα εργασία θα ήταν η χρήση σκαφών αναψυχής και ειδικά κάποια θέρετρα τα οποία θα προσφέρουν τέτοιες ε, υπηρεσίες για να καταπολεμηθεί ακριβώς αυτή η εποχικότητα του τουρισμού και να έχουμε τουρισμό όλο το χρόνο. Δεν ξέρω λοιπόν εάν η Κομισιόν θα μπορέσει να διαμορφώσει μια τέτοια πρόταση για να επαναληφθεί αυτό το μοντέλο και σε άλλα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Φώστερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Επίτροπο. Και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Φιντάντσα για το ότι πρόθεσε αυτό το θέμα, γιατί ο κύριος Χιγκίνης έχει δίκιο. Δεν το έχουμε συζητήσει και νομίζω πως ε, και εγώ έχω εργαστεί κάποια χρόνια στον τομέα του τουρισμού και τα κράτη-μέλη δεν εκτιμούν τα έσοδα που ε, υπάρχουν σε αυτόν τον τομέα, αν συνειδητοποιούν ε, τι γίνεται σε ολόκληρη την αλυσίδα με, μέχρι τον ταξιτζή που θα σε πάει στο ξενοδοχείο σου. Βεβαίω, το θέμα στον τουρισμό είναι πως ο ένας είναι ανταγωνιστής του άλλου εδώ μέσα, έτσι. Ο, κάθε χώρα προσφέρει διαφορετικό προϊόν και διαφορετικό πολιτισμό κτλ. Οπότε η ευθύνη είναι στη χώρα του καθενός μας για να κάνει ό,τι μπορεί σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για να ενθαρρύνουμε τον κόσμο από όλο τον κόσμο και την υπόλοιπη Ευρώπη να μας επισκεφτεί. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω πως σωστό είναι να εξετάζουμε ολόκληρο το προφίλ του τουρισμού, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό. Για το θέμα των θεωρήσεων βεβαίω μπορούμε να έχουμε mm. δυσκολίες δυσκολίε αν δεν υπάρχει αμοιβαιότητα. Δηλαδή, εμεί να διευκολύνουμε, αλλά όταν εμεί πηγαίνουμε από την Ιταλία και στην Ιταλία από το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μας διευκολύνουν τόσο. Ναι. Οπότε έχετε δίκιο. Δηλαδή πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικό το σύστημα. Να αναφερθώ τώρα και στην ποιότητα του προϊόντος. Δεν είναι εύκολο να τυποποιηθεί όλο το προϊόν, αλλά πρέπει να δώσουμε περισσότερο βάρος στο στην ε, αξία του προϊόντος, γιατί ο κόσμος δουλεύει σκληρά, πληρώνει τους ε, φόρους του και πάει διακοπές. Και δεν με ενδιαφέρει κάποιος ε, και δεν θέλω κιόλας κάποιος να χτίζει ένα ξενοδοχείο δίπλα σε αυτό στο οποίο μένω. Αλλιώς, αλλιώς δεν θα ξαναέρθω, ούτε θα το πω σε ένα φίλο μου. Επίσης τα προβλήματα που είχαμε με δηλητηρίαση μονοξιδίου του άνθρακα σε μια ασφαλή κτίρια και δεν μπορούμε βεβαίω να έχουμε τέτοια πράγματα στην Ευρώπη γιατί δημιουργούν άσχημη φήμη τα δυστυχήματα αυτά. Τώρα, κατά την άποψή μου, όταν έχουμε μεγάλα γεγονότα όπως η Ολυμπιακή Εμεί προφανώ στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαμε φανταστική χρονιά, είχαμε <laughs> και. Είναι επέτειο ανάληψη καθηκόντων της ε, Βασίλισσας, γιατί, για τη Βασίλισσα έρχονται να δουν έτσι, δεν έρχεται κανείς να δει τον Πρωθυπουργό, οπότε ε, και οι άλλες ε, χώρε που έχουν βασίλισσες ξέρουν τι εννοώ, οπότε πρέπει να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να έρθει και ε, νομίζω πως έχουμε ένα αρκετά καλό προϊόν. Ε, ναι, ε, έρχονται να δουν τη Βασίλισσα, ναι. Αυτά ε, θα έλεγα εγώ. Εμείς έχουμε ξανασυναντηθεί κύριε Επίτροπε στο Intergroup για τον εναερίο χώρο. Ναι. Λοιπόν, νομίζω θα συμφωνήσετε πως σημαντικό είναι να δούμε και τα, τις μεγάλες διοργανώσεις ποδόσφαιρο, κρίκετ, ό,τι είναι να έρχονται στην Ευρώπη, γιατί ακόμα και αν είναι ε, μια διοργάνωση στίβου, ξέρω εγώ, δύο εβδομάδων, δεν έχει σημασία, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, γενικά, νομίζω, αυτό το οποίο είπατε για τους Κινέζους, ναι, χρειαζόμαστε μεγαλύτερα αεροδρόμια και στις υποδομές μας για να έρχεται ο κόσμος. Ε, αυτή είναι μια ευθύνη που πρέπει να αναλάβουμε. Οπότε, έχω κάποιες ερωτήσεις για τον κύριο πίτροπο. Η πρώτη είναι, αναφέρατε τα 131 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολλά λεφτά. Ίσως να μην φαίνονται τόσα πολλά γενικότερα. Αλλά θα ήθελα να μάθω πού πηγαίνουν, γιατί προφανώς θέλουμε να ξοδευτούν σωστά. Δεν έχουμε κάποια αντίρρηση, αρκεί να προσθέτουν κάτι για να ωφεληθεί ο κλάδος. Και το δεύτερο ερώτημά μου είναι όταν άλλαξε η κυβέρνησή μας πριν από δύο χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, εγώ ήμουν με τον Υπουργό Τουρισμού σε μια διάσκεψη με όλους τους φορείς, αεροπορικές εταιρείε κτλ. για να δούμε τι θα γίνει με την πολιτική του κράτους για να βοηθήσει τον κλάδο μας. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, έχετε τακτικές συναντήσεις με τους υπουργού τουρισμού των κρατών μελών. Αν ναι, καλώς. Εάν όχι, γιατί όχι. Γιατί Θεωρώ πως οι Υπουργοί των κρατών μελών πρέπει να έρχονται στι Βρυξέλλες, να σε συναντάνε. Και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε νομίζω τις πληροφορίε που έχετε και τις πληροφορίε που έχουν οι Υπουργοί για να προχωρήσει αυτό το πρόγραμμα. Καλό κουράγιο λοιπόν. Ό,τι μπορείτε κάνετε, αλλά η ευθύνη είναι των κρατών μελών. Πρέπει λοιπόν να βρούμε διαδικασίες οι οποίες θα είναι απλές για να προωθεί αυτή η διαδικασία και να, είναι αρκετά ψηλά ως προτεραιότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε και προφανώς ευχαριστώ και τον κύριο Φιντάντσα. Ευχαριστώ κυρία Μπιλμπάου και μετά Μπενιόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Φιντάντσα και φυσικά και τον Αντιπρόεδρο Ταγιάννη για τις προσπάθειες που καταβάλουν ώστε ο τουρισμός πράγματι να είναι τομέας, τομέας που παράγει πλούτο, ε, κοινωνική ευημερία. Αυτό που είπατε για τις θεωρήσεις ε, με βρίσκει σύμφωνη, αυτό που είπατε επίσης ε, για το Ευρωπαϊκό Σήμα πρέπει να το προωθήσουμε. Το ζήτημα της εποχικότητας, συμφωνώ και κατάγομαι από τη χώρα των Βάσκων, που για συγκεκριμένες συνθήκες τα τελευταία χρόνια ε, δεν είχαμε την προτεραιότητα στον τουρισμό. Ε, ο πρώτος λόγος ήταν γιατί είμαστε εκβιομηχανισμένη περιοχή. Ναι, ναι, πράγματι. Έχουν πολύ μεγάλη βιομηχανική δραστηριότητα και μέχρι πρόσφατα είχαμε βέβαια και την τρομοκρατική οργάνωση ΕΤΑ ε, που είχε ως αποτέλεσμα να μην έρχεται σχεδόν κανείς να επισκεφθεί τη χώρα και αν κοίταζε προς τη χώρα των Βάσκων κοίταζε για να την αποφύγει πιο πολύ την περιοχή μας. Έχουμε τώρα όμως και τη μηχανική κρίση, αλλά ευτυχώς εδώ και κάποιο καιρό έχουμε την κατάπαυση πυρός από την ΕΤΑ. Ε, δεν έχουμε όμως πολύ ήλιο. Τέλος πάντων, η αλλαγή στην όλη κατάσταση έχει βοηθήσει να ε, προχωρήσει η χώρα των Βάσκων, το ΕΣΚΑΝΤΙ, και να βοηθήσει και ο τουρισμός στην οικονομική ανάπτυξη. Εγώ θα ήθελα να πω στον κύριο Ταγιάννη ότι νομίζω ότι υπάρχουν τρία θεμελιώδη πράγματα. Πρώτον, ορισμός ξεκάθαρων στόχων από ευρωπαϊκή σκοπιά. Επίσης, σαφής ηγεσία υπέρ του τουρισμού και τρίτον, επαρκής πόρη όπως ε, επιτράπει με τους σπόρους αυτούς πραγματικά να μετασχηματιστεί το Μπιλμπάο. Αντίστοιχα πρέπει να γίνουν προσπάθειες και πρέπει να δούμε τι προγράμματα, τι προϊόντα θα μπορούσαν να είναι ένας πόλος έλξης. Στη δική μας ε, περίπτωση είχαμε το Μουσείο Κούγκενχάιμ που πραγματικά εκτείναξε την ε, προσέλευση τουριστών ή ένα κέντρο προσέλευσης γαστριμαργικό με τον συνάδελφο Ουτζίας ε, ε, πήγαμε ε, και προσφέραμε τις εμπειρίες μας για το πώς μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκή καινοτομία και να γίνει ένα ποιοτικό άλλο στον τομέα της γαστρονομίας. Επίσης θα ήθελα να σας κάνω το εξής ερώτημα. Κάνατε προσπάθεια να αναλύσετε σε ευρωπαϊκό επίπεδο πέραν των ε, όλων προγραμμάτων που μας παρουσιάσατε, ποια είναι ε, τα βασικά στρατηγικά ε, προγράμματα, σημεία τα οποία θα μπορούσατε να πλασάρετε. Έχετε, να πείτε παραδείγματος χάρη στους αλλοδαπούς, έχετε πέντε λόγους για να έρθετε στην Ευρώπη. Π.χ. δεν έχετε μόνο το πύργο του Άιφελ για να πάτε στο Παρίσι ή το Μουσείο Γκουγκενχάιμ για να πάτε στο Μπιλμπάο, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα θέματα. Υπάρχουν, παραδείγματο χάρη, στο Μπιλμπάο πάρα πολύ ωραία μαγαζιά που πουλάνε κρασί και δεν είναι μόνο το Μουσείο Γκουγκενχάιμ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή μιλάμε για ποιότητα και συμφωνώ με το σήμα το ποιότητας Ευρώπη, αλλά δεν μιλήσατε για την εκπαίδευση. Όταν μιλάμε για ποιότητα, νομίζω ότι όταν κάποιος κοιτάζει προς την Ευρώπη και μιλάει για ένα ξενοδοχείο τριών, τεσσάρων, δύο αστέρων, σκέφτεται, πηγαίνοντας στην Ευρώπη, τι θα συναντήσω. Όχι μόνο τις υποδομές όμως, δεν εννοούμε αυτό μόνο. Ε, εννοεί ο τουρίστας πώς θα με υποδεχθούν εκεί, πώς θα με ε, προσέξουν, τι περιποίηση θα έχω. Και επομένως χρειάζεται και εκπαίδευση για να υπάρξει και μια εναρμόσει τέλο πάντων για να υπάρξει ποιότητα στην βερποίηση και στη φιλοξενία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εποχικότητα, ένα πιλωτικό πρόγραμμα νομίζω αναφέρατε ότι θα γίνει μια προσπάθεια με τη Βραζιλία, την Αργεντινή και τη Χιλή. Αν κατάλαβα καλά, θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί επιλέξετε αυτές τις χώρες ή απλά δώσατε ένα παράδειγμα. Και όταν μιλάμε για εποχικότητα και για πόρους, εγώ μιλώ για πόρους διότι εμείς στη χώρα των Βάσκων στις τρεις περιοχές μας, ε, όχι μόνο σήμερα, έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, που είναι η εξής. Επιδοτούνται ταξίδια ηλικιωμένων ε, ατόμων της τρίτης ηλικίας κάθε χρόνο υπάρχει ένα ειδικό πρόγραμμα ώστε αφενός να υπάρξει μια συνεργασία ε, στον τομέα το κοινωνικό και αφετέρου να, έχουμε το, να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της εποχικότητας ε, που πλήττει την Ισπανία αλλά και άλλες περιοχές της Ευρώπης. Θέλουμε λοιπόν να βρούμε, νέες, να βρούμε πρακτικές να, έχουμε, να προωθήσουμε το ποιοτικό σήμα και βέβαια υπάρχουν προγράμματα ε, πολύ καλά και παραδείγματα που αναφέρατε και εσείς, απλά θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θα κάνετε μια προσπάθεια για να εντοπίσετε καλές πρακτικές, γιατί έχουμε πολλά να σας προσφέρουμε εμείς από τη χώρα των Βάσκων. Ευχαριστώ. Λέω ο κύριος Μπενίν. Συμφωνώ με τους ομιλητές πως είναι καλό το ότι βλέπουμε με λίγο περισσότερη σοβαρότητα το θέμα. Έχουμε υποτιμήσει τον τουρισμό, δεν τον αντιμετωπίζουμε με τη σημασία που του αξίζει ως μέρος ευρωπαϊκής οικονομίας. Έτσι. Θα συμφωνήσω με την κυρία Μπιλμπάου πώς θα μπορούσαμε να προωθήσουμε κάποια θέματα στις νέες αγορές που αναφέρατε ε, οι οποίες ε, δεν είναι οι μόνες. Υπάρχουν και άλλες πιθανές δυνητικές αγορές για να έρθουν και άλλοι τουρίστες στην Ευρώπη. Στο έγγραφο αυτό του Brian Simpson και είχαμε μια εξαιρετική παρουσίαση πριν από λίγες εβδομάδες, αναφέρεται πως η Κομισιόν πρέπει να προωθήσει πιο έντονα τη βιομηχανική κληρονομιά της Ευρώπης, ε, η δυναμική της οποίας δεν έχει αναγνωριστεί και τονίζει πως ε, πρόκειται για ένα μεγάλο τομέα πολιτιστικού ενδιαφέροντος θα μπορούσε επίσης να ωφελήσει δευτερεύοντες προορισμούς και να οδηγήσει σε πιο μεγάλη διάχυση του τουρισμού στην Ευρώπη. Να ένα θέμα. Νομίζω πως το Ηνωμένο Βασίλειο βεβαίως ενδιαφέρεται κάπως περισσότερο από άλλες χώρες, αλλά έχουμε και στη χώρα μου βεβαίως μια ιστορική γέφυρα και στον Μπράιαν την περιφέρεια έχει παλιέ βιομηχανίε. Έχω πάει εγώ σε πολλά μέρη, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, που υπήρχε βιομηχανία. Και άλλα ανάλογα στη Γερμανία. Μπορούμε λοιπόν να φτιάξουμε ε, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Και νομίζω πως ε, υπάρχουν αρκετές δυνατότητες εδώ πέρα. Εγώ ούτω ή άλλω πολύ χρόνο σε γκαλερί, σε πινακοθήκε. και αυτά μπορούμε να τα δούμε. Δεν ξέρω λοιπόν τι κάνει η Κομισιόν αν τα σκέφτεται αυτά για να προωθεί την Ευρώπη και δεκτό είναι αυτό το οποίο λέει και η Τζάκη πως σε πολλέ περιπτώσει ο ένα ανταγωνίζεται τον άλλον. Αλλά μπορούμε να συνεργαστούμε για τις για τις ε, νεόπλητες αυτές περιοχές του κόσμου νομίζω για να προσελκύσουμε τουρίστες ε, στην Ευρώπη. Οπότε μπορούμε να αναπτύξουμε αυτά τα θέματα σε πανευρωπαϊκή βάση. Να αναφερθώ στις θεωρήσεις. Εμείς ε, και η Ιρλανδία δεν είμαστε στη Σέγγεν και εκεί πέρα να δείτε συζήτηση που γίνεται για το πόσου τουρίστες χάνουμε που πάνε στην υπόλοιπη Ευρώπη καθώς οι Κινέζοι έρχονται και πάνε σε πολλές χώρες της Ευρώπης με μια βίζα Σέγγεν, αλλά δεν ασχολούνται να βγάλουν και άλλη βίζα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν βλέπω λοιπόν πιθανότητα στο προσεχές μέλλον να μπούμε στη Σέγγεν, αλλά ελπίζω μακροπρόθεσμα. Εν τω μεταξύ υπάρχει κάποιος τρόπος να διευκολύνουμε μεταξύ Σέγγεν, Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας το πώς θα βγάζει κανείς τις δυο τρει βίζες αυτές μαζί σε ένα πακέτο. Ευχαριστώ, Ούτζο. Yeah, uh, so much, uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σου. Θέλω να πω ότι χάρηκα όλος ιδιαίτερος που είδα τα σημεία του εγγράφου, κυρίως το, τη δυνατότητα α, αναγέννηση που δημιουργεί ο τουρισμός. Και έτσι αυτή η αναγέννηση οδηγεί στην ε, παλινόρθωση των οικονομιών μας. Εκδόθηκε μια έκθεση πρόσφατα για το πιο εθνικό πάρκο α, ε, της ε, Βρετανίας, στην Νότια Αγγλία, στο Southtown, έχει μήκος 100 μίλια. Και λέει η έκθεση ότι του 465 εκατομμύρια το χρόνο ξοδεύουν οι τουρίστες. 8.200 θέσεις εργασίας. Προσέλκυσε 46 εκατομμύρια τουρίστες αυτό το πάρκο. Τι δείχνουν τα στοιχεία. Υπάρχει μεγάλο δυναμικό, πολλές δυνατότητες να αυξηθεί το χαμηλό ποσό που ξοδεύεται κατά κεφαλή. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε. Να εστιαστούμε επί μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται τα μοναδικά πράγματα που έχει να πουλήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολιτισμό, ιστορία, βιομηχανία, ε, φυσικό πλούτο, φυσική κληρονομιά. Είναι ιδιαίτερα ε, χαρακτηριστικά της Ευρώπης για τον οικολογικό τουρισμό. Μονοπάτια για ποδηλασία, όπως το διευρωπαϊκό δίκτυο συνδρομικό και το δίκτυο Eurovelo για τα ποδήλατα. Ε, πεζοπορία, με διαλύματα που μπορεί κανείς να χαλαρώσει και να εκπαιδευτεί σε πράγματα αναψυχής, όπως οι πιο ηλικιωμένοι. Τους αρέσει να βάφουν, να μαγειρεύουν, να ζωγραφίζουν. Ε, μικρής κλίμακας οι προσπάθειες, αλλά πρέπει να θαρρυνθεί ο κόσμος να περνά πιο πολύ χρόνο σαν τουρίστας, να απολαμβάνει αυτό που κάνει και να ξοδεύει χρήματα στην τόπια οικονομία. Άρα υπάρχουν τεράστιε δυνατότητε για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Σας παρακαλώ, κάντε ό,τι μπορείτε για να διευκολύνετε την ανάπτυξη σε αυτού του τομεί. Έτσι, κάποτε στο μέλλον, μπορώ να λέω σε αυτή την Επιτροπή ότι οι επισκέπτε που πήγαν στο Εθνικό Πάρκο του Staff Down, αυτά που δαπάνησαν οι επισκέπτε διπλασιάστηκαν ή τριπλασιάστηκαν. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, κυρία Γιάλα Σέντερ. <clears throat> Πρώτα είναι ο κύριος Ζούτζα, συγγνώμη. Ευχαριστώ, Κάρλο, ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Για την παρουσία σας εδώ και για την ε, παρουσίαση θα είμαι συνοπτικός. Δεν είναι εύκολο να μιλά κανείς στο τέλος. Να πω αμέσως ότι ξαναδιάβαζα το πρόγραμμα της ομάδας εργασίας, το έργο που έχουμε αναλάβει στην Επιτροπή και έχουμε πετύχει κάποια πράγματα, θετικός απολογισμός. Πρέπει να έχουμε επίγνωση του ότι ο χρονισμός είναι απαραίτητος όσον αφορά τον καθορισμό των στόχων. Ο χρόνος που περνά και οι στόχοι που δεν επιτυχάνονται καθιστούν τους ίδιους τους στόχους ε, ε, λιγότερο ε, χρήσιμους για το γενικό πρόγραμμα. Ξέρουμε ότι αυξάνεται η απασχόληση, αυξάνονται τα ποσοστά αν κάνουμε προσπάθειες. Πρέπει να αυξήσουμε όμως και την ταχύτητα υλοποίησης των προγραμμάτων ε, καθώς και των προτινωμένων μέτρων. Μετά από ένα χρόνο αυτό ήταν ενδιαφέρον να κάνουμε μια ανάλυση κύριε Επίτροπε. Να δούμε πώς ε, χρησιμοποιήθηκαν τα προτινόμενα χρήματα. Πώς προχωρούν τα πράγματα. Όσα μας αφορά, να δούμε πώς πηγαίνει η εφαρμογή της μεταρρύθμισης των στατιστικών στοιχείων για τον τουρισμό, κάτι που εγκρίναμε. Και δεν το χρησιμοποιούν όλοι αυτό. Δίνουν καμιά φορά στοιχεία, αλλά δεν το χρησιμοποιούν όπως θα έπρεπε. Εδώ και ένα μήνα, στην Ιταλία, στην οργάνωση BIT για τον τουρισμό, στην έκθεση, Κάποιες περιοχές είχαν στοιχεία του 2012 και οι περιφέρειες είχαν στοιχεία του 2010. Πώς μπορεί να εργαστεί κανείς και να κάνει προβλέψεις χρησιμοποιώντας στοιχεία τα οποία δεν είναι ε, πλέον χρήσιμα όσον αφορά τις προβλέψεις, για τις προβλέψεις. Δεν το καταλαβαίνω, ούτε μπορώ να φανταστώ ε, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, ο προγραμματισμός σωστά θα πρέπει πιο γρήγορα να προχωρήσουμε όσον αφορά την πραγματοποίηση των συζητήσεων των θεματικών. Εγώ είμαι διαθέσιμος να συμμετάσχω στη συζήτηση για την εποχικότητα και θέλω να κλείσω τη σύντομη παρέμβαση αναφερόμενο σε κάποια θέματα, κύριε Επίτροπε, που θα μπορούσαν να είναι και μια μικρή συνεισφορά στο σχέδιο αυτό το οποίο αναφέρατε. Εμείς χρειαζόμαστε εδώ να αποφασίσουμε σειρά διασυνδέσεων. Καθορίστηκαν ε, ε, ε, οι διασυνδέσεις λοιπόν που αφορούσαν διάφορες πτυχές, διάφορα θέματα. Δεν αφορούσαν μόνο τις μεταφορές. Δεν είναι μόνο αυτό. Επικοινωνία. Η δημιουργία ενός δικτύου προσφοράς. Επενδύσεις σε καινοτόμες υποδομές θα μπορούσε να δημιουργηθεί και μια πλατφόρμα για ανταλλαγή προσφοράς και ζήτησης εργασίας μεταξύ περιφερειών και χωρών που έχουν εποχικότητα εναλλακτική ή αντίθετη. Ε, έτσι θα εξασφαλίζεται συνέχεια στον αφορά την απασχόληση και την παραγωγή. Αυτό ισχύει για τα προϊόντα, για την εργασία, τις υπηρεσίες και για την επαγγελματική κατάρτιση διότι είναι πτυχές που μας ενδιαφέρουν. Και τέλος, Επίτροπε, νομίζω ότι το θέμα που ήδη εξετάσαμε, δηλαδή της εκόλαψης επιχειρήσεων, με στόχο να αφαιρεθεί η εποχικότητα σαν χαρακτηριστικό. Ίσως θα είναι ε, χρήσιμο εργαλείο για να βοηθήσει την υλοποίηση αυτού του προγράμματος, να υλοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό. Ε, Αγιάλα Σέντερ και μετά Κούν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας, για την προώθηση και ενεργοποίηση των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής για τον Τουρισμό. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Αντιπρόεδρο Ταγιάννη και να αναγνωρίσουμε ότι χάρη σε αυτόν τελικά φαίνεται να κερδίζει έτσι κάποια προβολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο τουρισμός γιατί είχαμε προβλήματα και κάποιες ατυχίες με τη δραστηριότητα αυτή που αποτελούν, αν θέλετε, στοιχείο ενεργητικού, περιουσιακό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή συζητούμε και το πολιετή προϋπολογισμό και πρέπει να δούμε πώς θα μπορούσαμε να το παρουσιάσουμε. Γιατί είμαστε υπέρ του να υπάρξει μεγαλύτερη ενίσχυση και πρόθεση του τουρισμού, γιατί είναι μια ευρωπαϊκή βιομηχανή σημαντική. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν πώς μπορεί να λειτουργήσει και ως ένας άξονας ε, κατά της κρίσης. Ε, οι χώρε που πλήττονται με σκληρότερο τρόπο από την κρίση είναι χώρε που εξαρτώνται και σε μεγάλο βαθμό την τουριστική δραστηριότητα. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη. Η κρίση επίση πλήττει και κάποιε ομάδε πληθυσμού, Οι ηλικιωμένοι, νέοι, οι άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, οι οικογένειε, οι μεσοαστικέ, οι χαμηλαστικέ, δεν ξέρω εγώ πώ θα τι ονομάσουμε. Το καλυψό επίση, το αρχικό το πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά προερχόταν από ένα γαλλικό, μια γαλλική δραστηριότητα και μια ισπανική δραστηριότητα, πώς θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε τα προγράμματα αυτά για να αντιμετωπίσουμε και την κρίση. Και σαν ενεργό πολιτική για την απασχόληση, για την καταπολέμηση της πώς μπορούμε να προωθήσουμε τον τουρισμό. Και επίσης θα μπορούσαμε να έχουμε επικαιροποιημένα και συνολικά στοιχεία για την προστέμενη αξία Δηλαδή, ταξιδεύουν ε, τα άτομα τη τρίτη ηλικία, ε, κάνουν τουρισμό. Εμείς στην Ισπανία βλέπουμε ότι μειώνονται δραστικά οι αριθμοί και λόγω υγεία κτλ. Επίση βλέπουμε κάπου να μην υπάρχει ε, τουρισμός, να σταματάνε οι δραστηριότητες αυτέ, και αυτό πλήττει και τι αεροπορικές ε, εταιρείε, για παράδειγμα. και πολλές άλλες επιχειρήσεις ε, που επηρεάζονται από, την τουριστική, από, τον, από τον τουρισμό. Οι ε, υπηρεσίες, ε, που παρέχουν υπηρεσίες ψυχαγωγίας, για παράδειγμα. Όλα αυτά πρέπει να τα εξηγήσουμε, να βρούμε τα κατάλληλα επιχειρήματα. Επίσης, πολιτική τουρισμού πάντα ως στοιχείο καταπολέμησης της κρίσης διατήρηση των ξενοδοχικών υποδομών και γενικότερα των τουριστικών υποδομών αυτό ουσιαστικά θα πρέπει να διατρέξει και τις άλλες πολιτικές, ενεργειακή απόδοση, δηλαδή ενεργειακά αποδοτικά κτίρια και ούτω καθεξής. Γιατί τα ξενοδοχεία, οι υποδομέ γενικά πολλέ φορέ αυτά δεν τα έχουν υπόψη του. Και θα πρέπει να δούμε πώ θα μπορούσαμε να προωθήσουμε μια, ένα είδο ε, τουριστικού εράσμου. Με το καλύψο υπήρχε η διάσταση αυτή αναφέρθηκαν κάποιες χώρες, ε, υπάρχουν και άλλες που δεν αναφέρθηκαν, όπως είναι η ΕΠΑ. Και σε ό,τι αφορά το σήμα το οποίο αναφέρατε, η Ένωση μέσα στην πολυμορφία είναι και το λογότυπο της ένωση. Πρέπει πράγματι να το προωθήσουμε. Έχουμε τις διαφορετικές παραδόσεις, ε, τη γαστρονομία, την υγεία. Πράγματι όλα αυτά μπορούμε να τα προωθήσουμε. Και στη δική μου περιφέρεια και στην Ευρώπη γενικότερα βλέπουμε ότι αναβιώνουν κάποιες ιστορικές δραστηριότητες. Ε, Παραδείγματο χάρη, αναβίωση κάποιου αγώνα, κάποιας μάχης ή κάποιου μεγάλου έρωτα, γίνονται κάποιε αναπαραστάσεις κτλ. Μήπως θα μπορούσαμε να επεξεργαστούμε και αυτό το θέμα σε βάθος και επίσης ε, για τις ίπα; ε, ξέρουμε ότι υπάρχει ιστορική σχέση Αμερικανών και Ευρωπαίων, πως και αυτό θα μπορούσαμε να το επεξεργαστούμε. Ευχαριστώ. Κάρλο, ευχαριστούμε και για την ε, πρωτοβουλία. Ήταν και ο Επίτροπο των Οικονομικών εδώ πέρα σήμερα. Τώρα, χωρί να αναφέρω συγκεκριμένου προορισμού, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια νούμερα. Το ΑΕΠ τη Ευρώπη με 500 εκατομμύρια είναι 12.000 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν ε, έχουμε το 5% που αντιστοιχεί στον τουρισμό είναι 600 δισεκατομμύρια ευρώ μιας μεσαίας χώρας μέλους. Τεράστιο ποσό, αλλά βεβαίως από την άλλη πρέπει να το σκεφτόμαστε και να λέμε τα λεφτά που δίνει ο κόσμος για τις διακοπές του τα έχουν ήδη βγάλει από κάπου αλλού. Έτσι. Οπότε όσο πιο δύσκολη είναι η κατάσταση, τόσο λιγότερα θα δίνουν για τον τουρισμό. Οπότε πρέπει γενικότερα η οικονομία να ανακάμψει στην Ευρώπη και τώρα ακριβώς πρέπει να σκεφτούμε σε ποιο προορισμό θα πάνε οι Ευρωπαίοι συμπολίτε μας. Τώρα εντάξει τα υπόλοιπα Ινδία, Σεϊχέλες, Αυστραλία και τα όλα αυτά τα λεφτά φεύγουν από τη δική μας οικονομία και πάνε εκεί πέρα. Στην Ευρώπη υπάρχουν όλοι οι προορισμοί που χρειάζεται κανείς. Κανένας Αμερικάνος δεν θα ερχόταν για σκι στην Ευρώπη ή για καταδύσεις ε, στην Ερυθρά. Μένουν όλοι στη χώρα τους. Και δίνουν τα λεφτά στη χώρα τους. Πρέπει και εμείς να το σκεφτούμε. Πού είναι η κοινή μας πρωτοβουλία. εντάξει το ε, outgoing, αλλά και εσωτερικά τι γίνεται. Νομίζω έχουμε να προσφέρουμε τα πάντα ε, και ιστορία και τα πάντα. Το, η, η, διεθνής, η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση τουρισμού είναι στο Βερολίνο και το σκέφτηκα. Η Ευρώπη δεν έχει ε, περίπτερο δικό της στην έκθεση αυτή. Να πει, ξέρω εγώ, συνολικά στην Ευρώπη κάνουμε διαφήμιση. Ο καθένας από εμά ξέρει τι γίνεται στη δικιά του χώρα και, ε, και εντός χώρας δηλαδή. Το ένα φέρετρο ανταγωνίζεται το άλλο. Αλλά να λέμε ότι έχουμε έναν προορισμό την Ευρώπη και όπου είναι κανείς να πάει, πάει. Νομίζω έτσι μπορούμε να προσθέσουμε προσθέμενη αξία, δηλαδή να μείνουν τα λεφτά εδώ στην Ευρώπη και να κάνουμε διακοπές εδώ. Ευχαριστούμε, Βέρνερ. Ευχαριστώ. Πού να συνοψίσει ο Αντιπρόεδρος. Έχει πάρα πολλά θέματα να συνοψίσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από αυτά που ετέθησα. Ευχαριστώ, Κάρλο. Πάνω απ' όλα, μία αξιολόγηση θα κάνω, Πολιτική φύσεως. Πιστεύω ότι από πλευρά όλων είδα ότι υπάρχει επίγνωση του πόσο σημαντικό είναι το βιομηχανικό τμήμα του τουρισμού ε, για την ε, ανάπτυξη της οικονομίας μας, για την αντιμετώπιση της κρίσεως και για προοπτικές που μπορούμε να δώσουμε στους νέους. Θεωρώ ότι η κοινή θεώρηση του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούσε να μας επιτρέψει να πετύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα από την πολιτική έποψη, όπως έλεγα, πριν από το τέλος της θητείας. Πριν τη λήξη της θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επίσης. Όπως υπενθύμιζε η κυρία Γιάλα Σέντερ, δεν ήταν εύκολο να θέσουμε στο επίκεντρο των συζητήσεων της βιομηχανικής πολιτικής στον τουρισμό. Το να λέμε στα διάφορα έγγραφα ότι ο τουρισμός είναι θεμελιώδης τομέας και για την επαναβιομηχανοποίηση της Ευρώπης, το να πείσει κανείς τα κράτη-μέλη που προβληματίζονται γιατί χάνουν τη συνέχεια ε, τις ικανότητές τους, τις δυνατότητες που έχουν, όπως και οι περιφέρειες που είχαν δυνατότητες. Και να μιλάμε για την ευρωπαϊκή πολιτική του τουρισμού. Στην αρχή υπήρχε δυσκολία να διοργανώσουμε ευρωπαϊκά συμβούλια που θα ασχολούνται με τον τουρισμό, να μαζεύονται οι υπουργοί. Απαντώ στην κυρία Φώστερ. Ναι, κάναμε διάφορες συνεδριάσεις. Ε, ενέπλεξα τους υπουργούς σε πολλές δράσεις, κοινέ δράσεις και υπογράμμισα τη συνεργασία με τους Υπουργούς Τουρισμού όσον αφορά την ανάπτυξη του προγράμματος του πιλωτικού των 50.000 τουριστών ε, με την Λατινική Αμερική. Γιατί Λατινική Αμερική. Διότι στη Λατινική Αμερική ζουν εκατομμύρια άτομα που έχουν καταγωγή Ισπανική, Ιταλική, Πορτογαλική, Γερμανική άτομα όπως υπεθύμιζε και ο όσον αφορά τους Ιρλανδούς ε, που έχουν ακόμα συγγενείς. Πιο φημισμένο παράδειγμα των τελευταίων ημερών είναι ο Πάπας, από την, ε, ο Αργεντίνος, που είναι, είχε ε, γονείς Ιταλούς. Και έγινε γιορτή στο χωριό καταγωγής των γονιών του. Και αυτό σε διασύνδεση με την Αργεντινή. Υπάρχουν σχέσεις με Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή. Πήγα στο Σαντιέγο τη Χιλή, πήγα σε αστιατόριο και είπα πόσο Γερμανοί ήταν η γιορτή γερμανική. Ήταν όλοι οι Αργεντίνοι που μιλούσαν γερμανικά, σαν μητρική γλώσσα μεταξύ του. Πραγματικότητα λοιπόν είναι αυτή που συνδέεται στενά με την Ευρώπη. Να τους πούμε, ελάτε κατά την ε, χαμηλή περίοδο να δείτε από πού προέρχεται η οικογένειά σας ή να ανακαλύψετε ξανά πού βρίσκονται οι συγγενείς σας. Είναι κάτι ή ελάτε να αγοράσετε και πράγματα που ε, είναι φτιαγμένα στο χωριό καταγωγή σου και πάρτα πίσω στην πατρίδα σου. Και η χρήση της γλώσσας βοηθά πολύ. Διότι είναι πιο εύκολο μετά να έχει κανείς τουρίστες που μιλάνε ευρωπαϊκές γλώσσες από ότι τουρίστες που μιλάνε άλλες γλώσσες. Υπογράψαμε τη συμφωνία λοιπόν με χώρε τη Ένωση που συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πιλωτικό αυτό πρόγραμμα που σα ανέφερα. Δεν θέλω να σταθώ μόνο στην Λατινική Αμερική με οι Ηνωμένε Πολιτείε, Ισραήλ. Υπάρχουν και άλλε χώρε με τι οποίε μπορούμε να συνεργαστούμε κάποιο ανάλογο πρόγραμμα από τη στιγμή που θα έχουμε θετικά αποτελέσματα από το πρόγραμμα αυτό. Θέλω, σαν στόχο, να προσελκύσω περισσότερου ευρωπαίου τουρίστε. Μάλλον έξω Ευρωπαίους, στην, Ευ... Ε, στην, ε, ε, τουρίστες εκτός Ευρώπης στην Ευρώπη και οι τουρίστε Ευρωπαίοι που, σε αντάλλαγμα των Ευρωπαίων τουριστών που πάνε εκτός Ευρώπης. Σίγουρα, εγώ θέλω να εργαστώ και για εσωτερικό τουρισμό. Προγράμματα για τους seniors, για την τρίτη ηλικία. Προγράμματα που ετοιμάζουμε. Το πρόγραμμα Καλυψό. Είναι όλα προγράμματα που έχουν σαν στόχο την αύξηση αυτή, του εσωτερικού τουρισμού. Προγράμματα που φορούν θεματικούς τομείς, όπως οι διαδρομές οι θρησκευτικές. Υπάρχουν τόσο άλλα τέτοια προγράμματα. Είναι πρωτοβουλίες που θέλουν να αναπτύξουν ε, τον τουρισμό εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως να προσθέσω και κάτι άλλο. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες του κυρίου Κουν. Έλεγε ας κάνουμε ταξιδέψουν τουρίστες μας στο εσωτερικό της Ευρώπης. Όμως για αυτό το πρόγραμμα ανταλλαγών που προανέφερα στη συμφωνία χρησιμοποιούνται οι αεροπορικές εταιρείες οι ευρωπαϊκές μόνο. Άρα το πρόγραμμα προβλέπει εκπτώσεις όταν ταξιδεύεις με ευρωπαϊκές εταιρείες όπως η Lufthansa. Ε, αυτό σημαίνει ότι κερδίζουν οι tour operators. Δεν είναι δεν θα πάνε και οι τουρίστες εξάλλου στο εξωτερικό, το λέμε εμείς. Τώρα όσον αφορά άλλο τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό των όσων έγιναν μάλλον. Από, στον κύριο Ούτζες απαντώ. Κάθε Φεβρουάριο στέλνω μια επιστολή κάπως πολυσέλιδη με όλες τις πρωτοβουλίες και τα επιτεθέντα αποτελέσματα. Όχι μόνο στον τομέα του τουρισμού, αλλά σε όλους τους τομείς αρμοδιότητάς μου, βιομηχανία, διάστημα, α, ε, τουρισμός. Βεβαίως θα γίνει μια αναθεώρηση ενδιάμεση ε, της δράσης που δρομολογούμε για την πολιτική του τουρισμού. Τα 21 περίφημα σημεία θα τα παρουσιάσω στο φόρουμ το ευρωπαϊκό στο Βίλνιους επί Προεδρίας στις 17 και 18 ε, Νοεμβρίου τρέχοντος έτους. Ε, απαντώ στον κύριο Χίγκη, στο ερώτημά σας όσον αφορά τις ημερομηνίε κλπ. Όπως όλοι οι Ιταλοί, στη, στη μητρική μας γλώσσα μιλάμε βιαστικά και γρήγορα και για τους φίλους μας τους διερμηνείς δεν είναι πάντα εύκολο να συνοψίζουν τα πάντα και να μεταφράζουν τα πάντα. Θα προσπαθήσω να μιλάω ίσως και λίγο πιο αργά. Είχα πει ότι η πρόταση κανονισμού για το ποιοτικό σήμα ή το σήμα ποιότητας Περιμένω να καθίσετε. Περιμένω να καθίσει. Λοιπόν, η πρόταση κανονισμού σχετικά με το σήμα ποιότητας, το ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας ήδη είναι στη φάση διαβουλεύσεων ε, σε διπηρεσιακό επίπεδο. Λοιπόν, ήδη είμαστε σε προθυμένο στάδιο και είναι θέμα εβδομάδων. Πιστεύω ότι σε τρεις-τέσσερις εβδομάδες, πριν από τον Ιούνιο, τουλάχιστον μεταξύ Απριλίου και Μαΐου, θα παρουσιάσω την πρόταση στους συναδέλφους μου και αμέσως μετά θα καταφτάσει στο Κοινοβούλιο. Ε, ελπίζω ήδη να έχουμε ένα αποτέλεσμα να έχει εγκριθεί σε πρώτη, να εγκριθεί σε πρώτη ανάγνωση από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο αυτή η πρώτη νομοθετική πρόταση. Πρώτη νομοθετική πρόταση για τον τομέα του τουρισμού που θα λέγαμε στον τουρίστα που έρχεται από μακριά και διατρέχει την Ευρώπη επί ένα μήνα, ταξιδεύει στην Ευρώπη για ένα μήνα, να του λέμε τι είδου ξενοδοχεία μπορεί να βρει τι τόπους μπορεί να επισκεφθεί. Για μας είναι πιο κοντινά όλα αυτά. Για εκείνους είναι άγνωστα πράγματα. Κινέζος ας πούμε. Έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Και σε κάποιο Ιαπωνέζο πρέπει να λέμε ποια είναι η ποιότητα. Αυτό το σήμα που θέλουμε να βάλουμε δεν, επουδενή δεν αντικαθιστά τα εθνικά σήματα. Είναι γενικό πλαίσιο που δίνει προστιθέμενη αξία, προστιθέμενη ποιότητα που μπορεί να παρουσιάζεται και να προβάλλεται στον κόσμο. Διαφορετικά έχουμε περιφερειακό σήμα, σήμα του ξενοδοχείου, εθνικό. Δεν μπορούμε να τη γινάμε στον κόσμο με 50 διαφορετικά σήματα ποιότητας διαφορετικά. Ένα ευρωπαϊκό σήμα ποιότητα εκπροσωπεί έναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή που αξιοποιεί κάποιους, ε, κάποιες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ξενοδοχεία που έχουν υψηλή ποιότητα. Όσον αφορά την πολιτική που θα πρέπει να εφαρμόσουμε, σίγουρα η οικονομική πτυχή είναι πάρα πολύ σημαντική. Καταφέραμε και στο Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κόπο. Δεν ήταν εύκολο να έχουμε στο κόσμο ένα κεφάλαιο που αφορά τον τουρισμό, διότι πολλοί επιμένανε και λέγανε ότι ισχύει επικουρικότητα, η αρχή της επικουρικότητας. Η αρχή της επικουρικότητας όμως, επιμένω, θεωρώ ότι είναι μία από τις βασικές αξίες της ένωσής μας. Όμως, το να έχουμε προστιθέμενη αξία δεν σημαίνει παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας, και να έχουμε ευρωπαϊκή πολιτική για την προώθηση της Ευρώπης στον κόσμο, για τη διαφήμιση της Ευρώπης στον κόσμο και για την ανάπτυξη εσωτερικού τουρισμού, να έχουμε τελικά ε, ε, θετικά αποτελέσματα οικονομικά, αυτό είναι σίγουρα σημαντικό. Όσον αφορά τη χρήση των πόρων, ο συνάδελφος Φιντάνς το υποστήριξε, ο αξιότιμος Φιντάνς τα χρήματα που χρησιμοποιούμε, τις πόρους που χρησιμοποιούμε. Ξεκινήσαμε το 2012 τη δημοσίευση διαγωνισμών για μελέτες για χαρτογράφηση, πλήρη χαρτογράφηση ζήτησης και προσφοράς απαιτήσεων για κατάρτιση σε θέματα προσβασιμότητας σε τουριστικές υπηρεσίες για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και ποιος είναι ο οικονομικός αντίκτυπος. Δημοσιεύθηκε και μια πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για τις προσπάθειες που έγιναν και την αριστεία που έχει επιτευχθεί για τον προσβάσιμο τουρισμό από πλευράς μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όσον αφορά αυτό το χρόνο έχουμε τέσσερις προτεραιότητες που, που αποτελούν, μάλλον βασίζονται από των αποτελεσμάτων. Θέλουμε καλύτερη συνεργασία με τους destination managers, με την τοπική αυτοδιοίκηση, θέλουμε να δημιουργηθούν δρομολόγια ε, αριστείας τουριστικά που να ε, αποτελούν εμπειρία και για τα άτομα με αναπηρία. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον πιο ευνοϊκό για την οθέτηση πρωτοβουλειών όσον αφορά το training, την κατάρτιση και κατάρτιση όσον αφορά τον τουριστικό τομέα, να χρησιμοποιηθούν εκτενέστερα οι καινοτομίε για το περιβάλλον, για προϊόντα και υπηρεσίες πιο βιώσιμα. Θα κάνουμε εξτατείες ενημέρωσης και ανακοινώσεις και θα οργανώσουμε εκδηλώσεις διαφημιστικές και σεμινάρια ad hoc Όλα αυτά με τα χρήματα τα οποία έχουμε λάβει. Όσον αφορά πάντα το σήμα ποιότητας, το είναι προστιθέμενη αξία, πιστεύω, όμως όσον αφορά το ερώτημα του κ. Ντεγκράντες, πάντα για τους σπόρους μιλάω, ξεκινήσαμε με την πρωτοβουλία Καλυψό το 2009 εντοπίσαμε τέσσερα, τέσσερις τομείς κλειδιά και δημιουργήθηκε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για να εντοπίσει και να γνωστοποιήσει τα ωφελήματα στις επενδύσεις στον κοινωνικό τουρισμό. Ε, δρομολογήσαμε μελέτη χαρτογράφηση τουριστικού τουρισμού σε 20 χώρες και δεσμευτήκαμε να διοργανώσουμε 7 εκδηλώσεις για την ευαισθητοποίηση των πολιτικών και του κοινού και να διευκολύνουμε και την συνάντηση των πλεκομένων. Διοργανώθηκαν στην, Πολωνία, Ρουμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Βέλιο αυτέ οι εκδηλώσει για να συναντηθούν όλοι αυτοί οι φορεί. Σαν αποτέλεσμα, ε, για τα φυλάδια και τι προσπάθειε που κάναμε για να διευκολύνουμε την ανταλλαγή τουριστών μεταξύ χωρών μελών, είχαμε σαν στόχο του εμπορευόμενου του τομέα. Χρηματοδοτούμε εννέα προγράμματα με 19 χώρε που συμμετέχουν. Αυτά τα προγράμματα μπορούν να οδηγήσουν στην πλατφόρμα Web Calypso που θα ξεκινήσει από τον Ιούνιο 2013. Συγχρηματοδοτείται από εμά και από τη Διεθνή Οργάνωση του Κοινωνικού Τουρισμού στα πλαίσια του προγράμματος TIP όπου εκείνοι που παρέχουν προσφορές για τον κοινωνικό τουρισμό και εκείνοι που θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις προσφορές μπορούν εύκολα να συναντηθούν. Το πρόγραμμα STIB θα ολοκληρωθεί το και μετά θα ακολουθήσει consortium για την πλατφόρμα Καλυψό και θα ξεκινήσει προσπάθεια με μία εκδήλωση, θα λάβει η χώρα στις Βρυξέλλες μέσα Μαΐου για αυτή την πλατφόρμα. Όσον αφορά τις πτυχές που πάντα συνδέονται με τους πόρους, τους διατιθέμενους, Περιμένω κάποιες πληροφορίες. Για το ερώτημα του κυρίου Δανέλη, όσον αφορά την παρά, τον παράκτιο τουρισμό, είναι ένα, ένας από τους 21 στόχους του σχεδίου δράσης μας. Ήδη συνεργαζόμαστε με την Επίτροπο, την κυρία Δαμανάκη, και ετοιμάζουμε μία ανακοίνωση όσον αφορά τον τομέα αυτό για να εφαρμοστεί αυτό το σημείο, να υλοποιηθεί. Και ανακοίνωση θα πρέπει να υιοθετηθεί ε, τον, Νοέμβριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά την οδηγία για τα πακέτα ταξιδιωτικά άλλα στοιχεία, δεν είναι αρμοδιότητά μου, της Επιτρόπου Ρέντινγκ, είναι, θα εγκριθεί, πιστεύω, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Βέβαια όλες οι ιδέες που δόθηκαν και ακούστηκαν την κυρία Γιάλα Σέντερ, Τεξέιρα κλπ. είναι πρόσδεκτα στοιχεία. Εδώ είναι οι υπάλληλοι της Γενικής μου Διεύθυνσης που ασχολούνται με τον τουρισμό. Όλες οι ιδέες που ακούστηκαν εδώ θα εξεταστούν και θα προσπαθήσουμε να τις εφαρμόσουμε. Όσον αφορά τους πιο μακρινούς τουριστικούς ε, προορισμούς Αζόρες και Μαδέιρα έγινε δελεχή συζήτηση στη συνέλευση της Δημοκρατίας εδώ και μερικές εβδομάδες όπου συνάντησα όχι μόνο τους βουλευτές αλλά και τη συνέλευση αυτών των δύο περιφερειακών προορισμών και τους κάλεσα να συναντηθούν με τη γενική μου διεύθυνση για να κουβεντιάσουμε. Θα προωθήσω και μια συνάντηση με στις γενικές διευθύνσεις που είναι αρμόδιες τα προβλήματα που έχουν οι περιφερειακές αυτές ε, ζώνες συμπεριλαμβανομένου και του τουρισμού εδώ στι Βρυξέλλε. Θα έχω φαντάζομαι ειδήσει από του εκπροσώπου των περιφερειακών αυτών ζωνών τη Μαδέιρα και των Αζωρών. Περιμένω ειδήσει για να μπορέσω να προχωρήσω. Η κυρία Φώστερ για τα στάνταρτ. Έχουμε ένα κανονισμό που ασχολείται με την ανάπτυξη προδιαγραφών ευρωπαϊκών τις προδιαγραφές και πρέπει να υπάρχουν πρότυπα και για τις υπηρεσίες. Τα, τα στάνταρ για τα προϊόντα περιέχουν και κάποια στοιχεία για τις υπηρεσίες και αντιστρόφως. Και τα στάνταρ για τις υπηρεσίες μπορούν να αφορούν και τα προϊόντα, να αναφερθούν στα προϊόντα. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορεί ο τουριστικό τομέα να τυποποιηθεί, να διερωτηθούμε. Βασίζεται σε εμπειρία, ο καθένα ζητά με τον τρόπο του τον τομέα αυτό και ζει αναλόγω. Μπορούμε να τυποποιήσουμε την ποιότητα μιας υπηρεσία. μπορούμε να τυποποιήσουμε την ικανοποίηση ενός τουρίστα. Δεν είναι εύκολο, όμως ε, πιστεύω ότι το σήμα της ποιότητα μπορεί και αυτό να είναι κάτι που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Όσον αφορά Α, ναι, την ευρωπαϊκή κληρονομιά. Αναφέρθηκε η πολιτισμική κληρονομιά, κυρίως η βιομηχανική κληρονομιά. Ξέρω ότι είναι ένα θέμα το οποίο αρέσει πολύ στον Brian Simpson. Είναι σημαντικά όλα τα προγράμματα και αυτό που αναπτύσσουμε με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο συμπεριλαμβάνει αυτό το τμήμα το πρόγραμμα αυτό που διαμορφώνεται από κοινού με το Συμβούλιο επικεντρώνεται επί τη ανάπτυξη εξαιτήτων των μάνατζερ που είναι επικεφαλή των πολιτισμικών διαδρομών, ενίσχυση τη κυβέρνηση των δικτύων τη Ευρώπη και τον περασμένο Δεκέμβριο ξεκινήσαμε τρίτο πρόγραμμα κοινή διαχείριση για να αναπτύξουμε και άλλο αυτέ τι δράσει που συμπεριλαμβάνουν διάδραση όλων των πολιτισμικών διαδρομών. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 12 μήνε με ένα προπολογισμό 500 εκατομμυρίων ευρώ και άλλο θέμα που ετέθη στη συζήτηση είναι της κατάρτισης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά δεν αφορά μόνο τον τουριστικό τομέα, είναι ένα θέμα που αφορά όλη την βιομηχανική πολιτική, το πρώτο σημείο του σχεδίου δράσης για την επιχειρηματικότητα αφορά αυτό μάλιστα, την κατάρτιση και προτείνω στα κράτη-μέλη, στα προγράμματα τα σχολικά, τον τελευταίο χρόνο του γυμνασίου να ε, έχει μαθήματα, προβλέπονται μαθήματα για το επιχειρήν, για το επιχειρηματικό πνεύμα, να εκπαιδεύονται οι νέοι να γίνουν ε, επιχειρηματίες ή manager. Αυτό γιατί, διότι στις χώρες όπου υπάρχει αυτού του είδους η κατάρτιση, η εκπαίδευση και με μαθητεία, στάζ, αυξάνεται ο αριθμό των νέων που γίνονται επιχειρηματίες ή μάνατζερ επιχείρησης. Η μανατζερ επιχειρηση εκπαίδευσης, κατάρτισης είναι θεμελιώδου σημασίας για όλους τους τομείς και ιδιαίτερω για τον τουρισμό. Γιατί επιμένω εγώ επί του τουρισμού σαν βιομηχανικό, σαν τομέας ε, σαν τομέα βιομηχανικό. Πέρασε η εποχή όπου υπήρχε το μικρό ξενοδοχείο με τη μαμά η οποία μαγείρευε για μας τη μακαρονάδα για τους Ιταλούς ή τάπα στην Ισπανία και ο πατέρας που παίρνει ε, κουβαλάει τις βαλίτσες και ο γιος μιλάει ε, με τα βίες κάποιες λέξεις αγγλικά και λοιπά και δεν υπάρχει ίντερνετ. Πρέπει να αλλάξει αυτό το μοντέλο εντελώς αν θέλουμε να είναι πραγματικά ανταγωνιστική στον κόσμο. Διότι στην Ανατολή, στην Τουρκία, στην Αφρική υπάρχει μια ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας της τουριστικής διοργάνωσης των επιχειρήσεων, που είναι πολύ ανταγωνιστικές. Εξάλλου, μία εκπαίδευση, μία κατάρτιση και διεθνοποίηση του τουριστικού μας τομέα, της τουριστικής μας βιομηχανίας, γίνεται θεμελιώδη σημασία. Κατάρτιση, ποιότητα, είναι και επισκεπτήρια που μπορούμε εμείς να παρουσιάζουμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σκέφτομαι πώς μπορεί να είναι καλό επισκεπτήριο ένα όμορφο ξενοδοχείο ευρωπαϊκό με Ευρωπαίους ε, καμαριε, καμαριαρίδες, με υπάλληλου Ευρωπαίους στη Σιγκαπούρη ή στο Πεκίνο όπου εκεί στο ξενοδοχείο πωλείται προϊόν υψηλής ποιότητας. Αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο θα ήθελα να το εξετάσουμε μαζί. Το έχω συζητήσει επανειλημμένα και με την ομάδα υψηλού επίπεδου που δημιουργήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη υψηλής μόδας ε, υψηλών προϊόντων. Όχι μόνο πασαρέλες, δεν μιλάμε για πασαρέλες και πράγματα μόνο για τους πλούσιους, είναι ένας τομέας που δίνει ε, σε χιλιάδες πάρα πολλούς ανθρώπους και πρέπει να χρησιμοποιηθεί που είναι δίδυμος τομέας με τον τουρισμό. Διότι όπου αυξάνεται ο τουρισμός, αυξάνεται και η πώληση αυτών των προϊόντων πολυτελείας. Αυτά τα προϊόντα είναι άριστο επισκεπτήριο στα άλλα μέρη του κόσμου. Αλλά όπως ξέρουμε, στην Κίνα, στην Ιαπωνία, τους αρέσει να αγοράζουν ε, το προϊόν και εκεί που παράγεται θα μπορούσαν ε, να αγοράζουν αυτό το προϊόν λοιπόν ε, ε, και στην Ευρώπη. Δεν βλέπει να βλέπουμε το προϊόν, τον τουρισμό σε έναν τομέα απομονωμένο, αλλά τομέα που συνδέεται στενά με πολλούς άλλους. Είμαι επιφεπισμένος όπως και η κυρία Φώστερ, ότι και μεγάλες εκδηλώσεις, το συμπεριλαμβάνουμε αυτό στη στατική μας του τουρισμό, οι μεγάλες εκδηλώσεις αποτελούν κατάλληλες στιγμές όχι μόνο για να προσελκύσουν τουρίστες απ' έξω από την Ευρώπη, αλλά να δημιουργήσουν ροές ε, ευρωπαϊκές ε, των τουριστών, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λονδίνου, η έκθεση Expo του Μιλάνου. Θυμηθείτε η Expo στην Κίνα, τι ήταν για την Κίνα και τι μπορεί να γίνει, όχι μόνο για το Μιλάνο, αλλά για κάποια πόλη τη Ιταλίας, αλλά για όλη την Ευρώπη, μία εκδήλωση Expo, μία έκθεση. Γι' αυτό Θέλει η Ευρώπη, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Μπαρόσο, θέλει να συμμετάσχει στη οργάνωση της έκθεσης του Μιλάνου, διότι μπορεί να γίνει αφετηρία έκθεση του Μιλάνου για αντίστοιχα γεγονότα στη Γερμανία, στην Αυστρία, στην Ουγγαρία, στην Ισπανία, έχοντας δύο διεθνή αεροδρόμια στο Μιλάνο. Και στην περιοχή να υπάρχουν διάφορα αεροδρόμια είναι πολύ εύκολο, πιο εύκολο να φτάσει κανείς ή να φύγει και να πάει σε άλλα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφωνώ να συναντήσω τη Βασίλισσα Ελισάβετ για την ώρα. Από τον Δούκα της Ιόρκης έχω προσκληθεί στο Buckingham για να συζητήσουμε για την πολιτική του διαστήματος. Αν η Βασίλισσα Ελισάβετ με καλέσει να μιλήσουμε για την τουριστική πολιτική, με τα χαράς να πάω για μία ακόμη φορά στο Buckingham για να ε, προωθήσω την, ε, τον τουρισμό στην Ευρώπη. Ε, σε αυτό το θέμα ε, συνήθως κακογλωσσ... μιλάνε άσχημα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν μιλήσαμε για την, ε, Ευρωπαϊκή, για την πολιτική, η Independent έγραψε δύο σελίδες και είπα στον Παρόζο, να, για, για το μόνο τομέα για τον οποίο λένε καλά λόγια στη Βρετανία, ε, για την Ευρώπη, είναι ο τουρισμός. Μόνο ο τουρισμός και το διάστημα είναι τομεί στου οποίου συνεννοούμεθα καλώ με τη Βρετανική κυβέρνηση. Απάντησα όχι σε όλε τι ερωτήσει, αλλά πέρασαν και πάνω από 20 λεπτά που προσπαθώ να απαντήσω. Η δική μου γενική διεύθυνση είναι πάντα στη διάθεσή σας όσον αφορά την πλατφόρμα ITC που ανέφερε νομίζω ο κύριος Δανέλης και ο κύριος Φιντάντσα ε, δημιουργήσαμε μια ομάδα εργασία στην οποία συμμετέχουν όλες οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις ε, του τομέα που συνεργάζονται μαζί μας για να επεξεργαστούν ένα πρόγραμμα που θα υποβληθεί και θα παρουσιαστεί μετά σε όλους τους ε, τουριστικούς φορείς. Λοιπόν, ο κύριος Κούν βλέπω ότι αναπηδά. Τώρα παπαντώ. Διοργανώνονται αποστολές μηχανικές για τη διεθνοποίηση. Πήγα και στο κολέγιο σας στην Πομερανία. Κάνει, έκανε πολύ κρύο και το βράδυ. Πολύ κρύο. Αλλά όμως φάγαμε πολύ καλά. Πο, πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες ε, τουριστικές τις συνοδεύουμε πηγαίνουν στην, ε, στον κόσμο. Κυρίως αποστολές για την κρίση γίνονται εντός, εντός Ευρώπης, όπως Ελλάδα, Πορτογαλία. Θα κάνουμε και κάποια αποστολή και στην Κύπρο και συνοδεύω και πολλές τουριστικές ε, επιχειρήσεις τις προάλλες στη Μόσχα επί τη ευκαιρία της συνάντησης με τον Υπουργό Πολιτισμού και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης που υπέφερε τον τουρισμό συναντήθηκα και μου ζητήθηκε να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας της Ευρώπης φορείς δηλαδή που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και διοργάνωσης διότι έχουν πολλούς πόρους αυτοί, αλλά χρειάζονται επιχειρηματίες που μπορούν να διοργανώσουν, ξέρουν να διοργανώνουν δραστηριότητες τουριστικές. Συνοδεύσαμε και στην Αίγυπτο επί τη ευκαιρία της Μεγάλης Αποστολής για την Ανάπτυξη 100 επιχειρήσεις τουριστικές ευρωπαϊκής σε μια συμφωνία με την είπα το εκπρόσωπο αντιπρόεδρο Άστον και θες, θέλαμε να προωθήσουμε τον τουρισμό μέσω κοινοπραξιών joint venture που αφορούν και τις κρουαζιέρες Διότι θεωρήσαμε όταν θα ηρεμήσει κατά στη Βόρεια Αφρική η πτυχή των κρουαζιερών μπορεί να είναι σημαντικό κομμάτι συνεργασίας διότι ήθελα να αποφύγω άμα ηρεμήσει η κατάσταση στη Βόρεια Αφρική οι τουρίστες που εμείς κατακτήσαμε και αποκτήσαμε διότι φοβόταν να πάνε στη Βόρεια Αφρική να μην έρχονται πλέον στην Ευρώπη και, να, και και να πηγαίνουν αλλού. Άρα η κρουαζιέρα στην περιοχή της Μεσογείου μπορεί να αντιπροσωπεύει ιδεώδη κοινοπραξία, joint venture μεταξύ ε, Μεσογείου και Βορείου Αφρικής ε, για να αυξηθεί ο τουρισμός και να μην χάσουμε σημαντικό κομμάτι ε, τουριστικό που έχουμε αποκτήσει αφού ηρεμήσει η κατάσταση και να μην ξανάρχονται στην Ευρώπη. Το ίδιο ισχύει και για τις τουριστικές κρουαζιέρες στη Βόρεια Ευρώπη, θάλασσα Μπάρεντς, Νορβηγία κλπ. Ε, και εκεί θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμεθα. Είμαι πάντα στη διάθεσή σας για οδήποτε ερώτημα, ε, ό,τι χρειαστείτε ό,τι χρειαστεί το Κοινοβούλιο, ό,τι θεωρεί σημαντικό το Κοινοβούλιο, για να προσπαθήσω να σα δώσω όσο πιο γρήγορα μπορώ απαντήσει. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή, ευχαριστώ για τι ερωτήσει και για τι ιδέε. Ελπίζω να υπήρξα επαρκώ σαφή. Ευχαριστώ, Αντιπρόεδρε, για το εύρο των απαντήσεων που δώσατε. Αν υπάρξουν ερωτήσεις για λεπτομέρειες, αν ερωτήσεις δεν πήραν κάποια σαφή απάντηση, βεβαίως μπορείτε άμεσα να απευθυνθείτε στις υπηρεσίες του Αντιπροέδρου και τον ευχαριστώ που είναι πάντα διαθέσιμος. Συμφωνείτε Αντιπρόεδρε να ζητήσετε τις υπηρεσίες σας να μας δώσετε, να δώσετε κάποιες απαντήσεις και τη σχετική τεκμηρίωση και να δώσετε τα έγγραφα στην γραμματεία μας, διότι δεν καταλάβαμε ίσως κάποιες από από απαντήσεις. Λοιπόν, θα δώσω την Προεδρία. Δέχομαι την πρόσκλησή σας να εμβαθύνουμε σε αυτό που κάναμε, στο έργο που κάναμε στατιστικές και στην επικαιροποίηση του κανονισμού για τα στατιστικά για τον τουρισμό που εγκρίθηκε εδώ και δύο χρόνια. Όσον αφορά τις, ε, το πώς λειτουργεί το Task Force, η ομάδα εργασίας, ο πρόεδρος Σίμψος στην αρχή της συνεδρίασης είχε προβλέψει ότι μετά αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα θα δούμε πώς θα κινηθούμε, τι θα κάνουμε. Μην πεπισμένους ότι πρέπει να προωθήσουμε αυτά τα θεματικά, θεματικές συζητήσεις με τη συμμετοχή των stakeholders και των μελών της Task Force. Λοιπόν, μπορεί να, όποτε θέλετε, είσαστε και φιλοξενούμενο και δικός μας και τη Επιτροπής Τουρισμού. Χρειάζεται μια task force για να επεξεργάζεται λεπτομέρειες με τη συμμετοχή αυτών που ε, συζητούν στο task force. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε αυτά με τον ε, πρόεδρο Σίμψον μετά την διακοπή των, του Πάσχα. Λοιπόν, καλό Πάσχα σε όλους και καλό βράδυ. Γεια σας.